Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Το πρώτο σημείο στη διάταξη είναι η δήλωση της Επιτροπής, δηλαδή προτινόμενη οδηγία περί προστασίας των δεδομένων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυχάνουν χάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικέ υποθέσεις. Θα ήθελα να επιθυμήσω στα μέλη ότι σε αυτή τη συζήτηση δεν προβλέπεται διαδικασία catch the eye. Η Επίτροπος κυρία Μαρία Δαμανάκη έχει το λόγο εξ ονόματος της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Dear President, dear colleague... Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Επιτροπή κατέθεσε τις προτάσεις μεταρρύθμισης ε, για το Ευρωπαϊκό Καθεστώς Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τον Ιανουάριο για δύο λόγους. Καταρχάς για να εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων για ε, ιδιώτες όπως προβλέπετε, για τους ιδιώτες όπως προβλέπετε στις συνθήκες και δεύτερον για να προσφέρει σε ευρωπαϊκές υπηρεσίες ε, ένα ουδέτερο αλλά και ασφαλές σύστημα προστασία των δεδομένων για το μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να προχωρήσουμε ταχαίως προς την επίτευξη συμφωνίας για τη δέσμη μέτρων που έχει τεθεί επιτάπητος. Το Κοινοβούλιο έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στα έγγραφα εργασίας και στα σχέδια εκθέσεων που προετοίμασαν οι εισηγητές. Για δε την Επιτροπή πρόοδος σημαίνει ο κανονισμός και η οδηγία να συνεχίσουν να ε, τη χάνουν διαπραγματεύσεως ως σύνολο ενιαίο. Γιατί το μέλλον και η ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών είναι οι δύο όψει του ίδιου νομίματο. Έχουμε να κάνουμε δύο πτυχέ τη πολιτική που θα επιτευχθούν χάρη στην υιοθέτηση, εφόσον γίνει αυτή, των προτάσεων για τη μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών κανόνων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που την χάνουν επεξεργασία στο πλαίσιο τη αστυνομική και δικαστική συνεργασία. Έχουμε ενισχύει μια πληθώρα ε, νομοθετημάτων και κανόνων. Η θέση ενισχύ της συνθήκης ε, της Λισαβόνας επιτρέπει την θέσπιση ενός ευρέως φάσματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ενός πλαισίου ευρέως, με προστασία των προσωπικών δεδομένων για τους ιδιώτες, ενώ ταυτόχρονα θα γίνεται σεβαστή και η ιδιαίτερη φύση της ε, αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας στα θέματα ποινικού δικαίου. Ιδιαίτερα, ιδιαίτερα ή το αναθωριωμένο πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να καλύψει πλέον και την ενσωτερική αλλά και τη διασυνοριακή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με περιορισμό έτσι των διαφορών ε, σε επίπεδο νομοθεσιών των κρατών μελών. Το status quo δεν διευκολύνει πάντοτε την απρόσκοπτη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών. Η το σύνολο των κανόνων, οι διατάξεις που ισχύουν και ίσιαν πριν από την συνθήκη της Λισαβόνας και που στόχο έχουμε τώρα να αναθεωρήσουμε, περιορίζουν την ε, δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων σε υπερσυνεριακό επίπεδο. Έτσι λοιπόν μπορεί να μην έχουν πάντοτε τη δυνατότητα οι αστυνομικέ και δικαστικές αρχές τη δυνατότητα να διακρίνουν μεταξύ της διασυνοριακής, της εσωτερικής επεξεργασίας των δεδομένων και δεν είναι πάντοτε εφικτό να γίνει η διάκριση στο, στην καθημερινή εργασία είτε του αστυνομικού είτε του δικαστηρίου. Επί παραδείγματι, μια ενιαία βάση δεδομένων, εθνική, που μπορεί να αξιοποιείται για την επιβολή του νόμου, μπορεί να περιλαμβάνει δεδομένα που έχουν συλλεγεί σε επίπεδο εθνικό ή που έχουν αποσταλεί από ε, άλλο κράτος μέλος. Έτσι λοιπόν θα ήταν μη αποτελεσματικό το να δημιουργηθούν δύο χωριστές ε, βάσεις δεδομένων σε τέτοιες περιπτώσεις, σε τέτοιες υποθέσεις. Επίσης θα ήταν μη αποδοτικό και εφαρμόσιμο το να εφαρμόζονται δύο διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες προστασίας για μία και μόνη βάση δεδομένων, ανάλογα με την προέλευση των δεδομένων αυτών. Έτσι λοιπόν, η προτινόμενη οδηγία στόχο έχει να καλύψει τόσο τα ε, εσωτερική συλλογή όσο και τα διασυνοριακή προελεύσεω δεδομένα, όπω άλλωστε είχε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η προτινόμενη οδηγία επίση περιλαμβάνει τη, καλύπτει τις ίδιες αρχές προστασίας με αυτές που έχουν εγγραφεί στον κανονισμό αντικατοπτρίζοντα έτσι πάλι το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επέκταση της ε, εφαρμογή των ε, κανόνων γενικής προστασίας, στου τομείς της αστυνομία και τη δικαστική συνεργασία. Κέρια στοιχεία για που έχουν εγγραφεί στο σχέδιο του κανονισμού συμπεριλαμβάνονται και στην προτινόμενη οδηγία. Επί παραδείγματι, η προστασία των δεδομένων ε, καταρχήν η προστασία, η σημασία του ε, αξιωματούχου προστασίας, η υποχρέωση κοινοποίησης και ανακοίνωσης τυχών παραβάσεων και η δυνατότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λαμβάνει, δυνα... να λαμβάνει αποφάσεις προσαρμογής σε σχέση με αποφάσεις τρίτων κρατών. Έτσι υπογραμμίζεται η σημασία μιας στεναρής, μιας στέρης προστασίας των προσωπικών δεδομένων και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε το γεγονό ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί δικαίωμα εγγεγραμμένο στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Γι' αυτό οι νέε αυτέ διατάξει για την προστασία των δεδομένων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και στα τομεακά νομοθετήματα, ιδιαίτερα στον τομέα του λεγόμενου πρώην του πυλώνα και άπαξ και τεθεί σε εφαρμογή η σχετική νομοθεσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει τρία χρόνια περιθώριο για να, μέσα σε τρία χρόνια μάλλον, θα πρέπει να αναθεωρήσει και ενδεχομένω να τροποποιήσει άλλα νομοθετήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία ενδεχομένω ρυθμίζουν την επεξεργασία των ε, προσωπικών δεδομένων από τι αρχέ ε, επιβολή του νόμου. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Επίτροπε, now speakers on behalf of the political groups. I call Mr. Καλό τον κύριο Κέλλη εκ μέρου των πολιτικών ομάδων και συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που μου δίνετε δύο λεπτά να μιλήσω για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Ένα σημαντικό θέμα για κάθε πολίτη, για κάθε επιχείρηση. Και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε όλο τον κόσμο είχαμε μια οδηγία ε, για την προστασία των δεδομένων που ήταν συναφής και μέρος αυτής της οδηγίας ε, είχε να κάνει με την επεξεργασία προσωπικών ε, δεδομένων από την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές. Αυτό ήταν το πλαίσιο, ήταν μια απόφαση πλαίσιο. Με τον χρόνο το Ευρωκοινοβούλιο συνειδητοποίησε ότι ήταν παροχημένη και ζήτησε την αναθεώρηση στην πραγματικότητα δεν ήταν ε, αποτελεσματική από διάφορες απόψεις, διότι είχε να κάνει με τη διασυνοριακή επεξεργασία, αλλά όχι σε εθνικό επίπεδο από την αστυνομία και ε, είχε ε, ευρείες ερμηνείε σε κρατικό επίπεδο και κάποια κράτη-μέλη είχαν υψηλά πρότυπα προστασία προσωπικών δεδομένων και άλλα χαμηλά. Και βέβαια η Επιτροπή είχε τις δικής της του ε, κανόνες. Και όπως είπε και η Επίτροπος, με την συνθήκη της Λισαβόνας και την εξέλιξη του διαδικτύου και τον μεταβάλλομενο κόσμο, χρειάστηκε επικαιροποίηση. Το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο θα προτιμούσε ένα ενιαίο μέσο ε, και, αλλά μπορούμε να δεχτούμε την πρόταση της Κομισιόν, ένα κανονισμό και μια οδηγία. Όμως μας ανησυχούν κάποιες πτυχές, ιδιαίτερα σε σχέση με την έλψη του επιτακτικού σε επίπεδο Συμβουλίου να ασχοληθούν με την οδηγία. Υπάρχει κάποια κίνηση στο επίπεδο του κανονισμού, αλλά όχι αρκετή στο επίπεδο τη οδηγία. Και γι' αυτό το λόγο θα ζητήσουμε από το Συμβούλιο να προωθήσει ένα δικό χάρτη για το πώ ε, θα προχωρήσουν και επίση να διασφαλίσουν ευελιξία σε ε, επίπεδο κράτου μέλου. Να μην υπάρχει ε, υπερβολικά ψηλά επίπεδα σε ένα κράτο μέλο και χαμηλά σε άλλο. Και, και τελικό σημείο και χαίρομαι να αναφέρω ότι ο Ιρλανδός Πρωθυπουργό ε, με προσέγγισε την περασμένη εβδομάδα και είπε ότι κατά τη διάρκεια της Ιρλανδική προθεσμίας θα το θέσουν ως μία από τις προτεραιότητές του. Σας ευχαριστώ. Ε, κύριε Κέλλη, η κυρία Τικάου θέλει να κάνει χρήση της ε, μπλε κάρτας. Κύριε Κέλλη, η κυρία Τικάου θέλει να κάνει χρήση της μπλε κάρτας. Αποδέχεστε το αίτημα της κυρίας Τικάου. Κυρία Τικάου, έχει το λόγο. Σύντομα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κέλλη αν ε, στον ε, φίλο πορεία που περιμένει από το Συμβούλιο θα ζητήσει να καταχωρηθεί και το ακόλουθο σημείο. Ο τρόπος με τον οποίο το νέο πακέτο θα επηρεάσει τις ε, διεθνείς συμφωνίες όπως SWIFT ή ε, το, την καταχώρηση των ονομάτων των επιβατών. Θα πρέπει να ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι συμφωνίες θα ευθυγραμμιστούν με το νέο πακέτο σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Yes, I think that's uh, very important. Ναι, νομίζω είναι σημαντικό αυτό το σημείο, διότι θα πρέπει να υπάρχει ε, συνέπεια σε όλα. Μπορώ να προβλέψω τι θα κάνει το Συμβούλιο, αλλά είναι σημαντικό να λάβουν όλα αυτά τα σημεία υπόψη τους και ιδιαίτερα ε, να ε, κινηθούν πιο γρήγορα στο θέμα αυτό, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αυτή της εντολής. Ε, και αν δεν ε, ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος ε, του επόμενου χρόνου με τις επικείμενες εκλογές το 2014 θα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί πρόοδος αν μένουν πολλά να γίνουν μέσα στο 2014. Σας ευχαριστώ. Δρόμο της ομάδος S&D, το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Δημήτριος Δρούτσας για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πάρα πολύ και την κυρία Επίτροπο για την παρουσία της εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την σημερινή δήλωσή της. Νομίζω λέω το αυτονόητο και συμφωνούμε όλοι μας σε αυτό ότι το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της Ευρώπης είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας, απαιτεί από όλου μας την δέουσα σοβαρότητα και προσοχή και να τονίσω για άλλη μια φορά ότι εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδίδουμε ακριβώ αυτή τη μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα. Και για ακριβώ αυτόν τον λόγο το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο είναι και θα συνεχίσει να είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και αυστηρό απέναντι στους υπόλοιπους θεσμούς της ένωσής μας σε αυτό το θέμα. όπως σας είναι γνωστό κυρία επίτροπε το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο επιθυμούσε από την αρχή ένα και μοναδικό νομοθετικό εργαλείο έναν κανονισμό που θα κάλυπτε όλες τις πτυχές και όλους τους τομείς που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων ώστε να αντιμετωπίζεται ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας ισότιμα παράλληλα δεν να συμπεριληφθούν και περιπτώσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές. η επιθυμία μας αυτή δυστυχώς ε, δεν έγινε σεβαστή με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε να διαχειριστούμε τις προτάσεις για έναν κανονισμό και μια οδηγία. παρ' όλα αυτά όμως το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο καλωσόρισε τις προτάσεις της επιτροπής αποφασίσαμε όμως να τις θεωρήσουμε και να τις αντιμετωπίσουμε ως ένα ενιαίο νομοθετικό πακέτο σε πρακτικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο ουσίας. για εμάς και θα ήθελα να το τονίσω αυτό δεν μπορεί να υπάρξει κανονισμός χωρίς οδηγία και θα επιμείνουμε στη λογική του πακέτου προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή και η ασφάλεια δικαίου. και χαίρομαι κυρία επίτροπε που και σήμερα με την παρέμβασή σας επιβεβαιώσατε για άλλη μια φορά ότι και η επιτροπή βλέπει και αντιμετωπίζει κανονισμό και οδηγία ως ένα πακέτο. Κύριε Επίτροπε, από την Επιτροπή, πιστέψτε με, δεν έχουμε παράπονα. Αντιθέτως, η συνεργασία με την Επιτροπή είναι σε εξαιρετικό επίπεδο και δεν διστάζω να το τονίσω αυτό από αυτό το βήμα και να σας εκφράσω και τις ευχαριστίες μου γι' αυτό. Δυστυχώς, δεν μπορώ να πω το ίδιο και για το συμβούλιο και ρωτώ πού είναι σήμερα το συμβούλιο σε αυτή τη συζήτηση γιατί δεν βρίσκεται σήμερα εδώ να απαντήσει σε σχετική προφορική ερώτηση που του θέσαμε. και επιτρέψτε μου να πω ότι πέρα από ένδειξη ασέβειας απέναντι στο θεσμό του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου αναγκάζομαι να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι το συμβούλιο δεν αποδίδει την απαραίτητη σημασία σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα για τους ευρωπαίους πολίτες δυστυχώς το συμβούλιο καθυστερεί τις εργασίες του για την οδηγία και αναρωτιέμαι και νομίζω εύλογα για ποιον λόγο το συμβούλιο με τη στάση του αυτή αρνείται να συνεργαστεί. επιτρέψτε μου κύριε πρόεδρε να ολοκληρώσω τονίζοντας ότι το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο θα υπερασπιστεί τις θέσεις του με κάθε μέσο που κρίνει απαραίτητο και κατάλληλο ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να τεθούν σε εφαρμογή ο κανονισμός και η οδηγία ως πακέτο παρέχοντας στους ευρωπαίους πολίτες υψηλού επίπεδου προστασία των προσωπικών δεδομένων τους. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ να κρατάτε στο ελάχιστο τη διάρκεια των παρεμβάσεών σας. Ο έχει συνάδελφος κυρία Σοφία Yes, thank you, Chair. Um... Μικρόφωνο, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για όσους από εσά παρακολουθείτε τις ε, προεδρικές εκλογές ε, στις Ηνωμένες θα ξέρετε για τι πράγμα μιλάω. Ε, ε αισθάνομαι λιγάκι σαν τον κλείδι Ίσχου μιλώντας απέναντι σε μια διακαρέκλα, γιατί ακόμα μια φορά απουσιάζει το Συμβούλιο. Οι συνάδελφοί μου ήδη υπογράμμισαν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επιμείνει στην ε, προσέγγιση τη συνολική. Δηλαδή ότι θέλουμε να είναι πακέτο ε, ο κανονισμός και η οδηγία. Θέλω όμως να προσθέσω κάτι, ότι η οδηγία για μας είναι προϋπόθεση για την περαιτέρω συνεργασία την αστυνομική και δικαστική. Γι' αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το καταλάβει το Συμβούλιο. Γιατί και το Συμβούλιο θέλει επιθυμίες και αυτό θέλει να προχωρήσει. Όπως και εμείς στον τομέα της ε, ε, αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας. Πώς μπορούν όμως αυτοί να ανταλλάξουν στοιχεία αν δεν υπάρχει επαρκής προστασία των δεδομένων. Γι' αυτό λοιπόν θα παρότρινα το απόν Συμβούλιο ε, θερμά να προχωρήσει γρήγορα με την οδηγία. Και θα ήθελα ε, να πω στους συναδέλφους, δεν θέλουμε roadmap, θέλουμε αποτέλεσμα, για γρήγορο αποτέλεσμα. Αν το Συμβούλιο θέλει να ενδυθούν περαιτέρω μέτρα στον τομέα της συνεργασίας, αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, μπορώ να σκεφτώ διάφορα ε, ενδιαφέροντα θέματα, ένταλμα ανάκρισης ε, κλπ. Αλλά επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω στο Συμβούλιο ότι ο, ο προκάτοχος αυτής της οδηγίας, η, η απόφαση πλαίσιο δηλαδή που ισχύει σήμερα, καταψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο. Ε, δυστυχώς αυτό έγινε πριν από τη Λισαβόνα, αλλά δεν θεωρούμε ότι η παρούσα ε, απόφαση πλαίσιο είναι επαρκής. Ό,τι και θα να κάνει λοιπόν το Συμβούλιο και ό,τι και να προτείνει θα πρέπει να είναι αρκετά καλύτερο από αυτό που ισχύει σήμερα. Δεύτερον, εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να ευθυγραμμιστεί η οδηγία με τον κανονισμό. Γιατί είμαστε απογοητευμένοι που υπάρχουν δύο νομικά μέσα και όχι ένα. Θα εργαστούμε λοιπόν και θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ σκληρά ούτως ώστε να έχουμε ένα εναρμονισμένο ενιαίο επίπεδο προστασίας δεδομένων για οποιαδήποτε χρήση ε, των δεδομένων αυτών, των προσωπικών δεδομένων. Και τέλος, συνάδελφοι, ε, για να επανέλθω στην αναφορά μου στον Clint Eastwood, ήθελα να πω το εξή στο Συμβούλιο. Όπως είπε ο Clint Eastwood όταν έπαιζε το ρόλο του Dirty Harry, όταν ένας ε, εγκληματίας τον αμφισβητούσε και τον προκαλούσε, του είπε κάνε στον, εαυτό σου ε, μία ε, ε, ερώτηση. Αισθάνομαι τυχερό. Έτσι θα πρέπει και το Κοινοβούλιο να προκαλέσει το Συμβούλιο. Και τώρα δίνω το λόγο στον συνάδελφο κύριο Άλμπρεχτ. Εκ μέρου των Πρασίνων. Ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε συζητούμε εδώ και σήμερα όχι μόνο την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά το μέλλον της συνεργασίας των αστυνομικών και δικαστικών αρχών στην Ευρώπη. Εδώ και χρόνια οι Υπουργοί των Εσωτερικών ε, προωθούν την ε, συνεργασία μεταξύ δικαστικών και αστυνομικών αρχών που είναι και απαραίτητη πρέπει να πούμε αλλά επαρελειμμένο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προειδοποιεί ότι οι κοινέ προδιαγραφές για την προστασία του κράτους των ε, συνόρων κτλ. Δεν, μπορούν, δεν μπορεί να παραγνωρίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για άλλη μια φορά όμως αυτή η απέτηση παραγνωρίζεται από το Συμβούλιο και ενώ αναγνωρίζονται τα αστυνομικά μέσα και μέτρα ε, παραγνωρίζετε το γεγονό ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές ω προ τι προδιαγραφές επιβολής του νόμου μεταξύ των κρατών μελών και ιδιαίτερω όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η υφιστάμενη λοιπόν ε, οδηγία ε, τώρα προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτές τις διαφορές χωρίς να κερδίζουν πολλά σε δικαιώματα οι εμπλεκόμενοι, τουλάχιστον το race to the bottom, δηλαδή ο αγώνας δρόμου προς τα κάτω, ως προς τις, ε, στην τήρηση των προδιαγραφών από τις αστυνομικέ αρχές, μάλλον θα σταματήσει. Και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να περιορίσουμε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Ωστόσο, το Συμβούλιο των ε, Υπουργών δεν, δεν δείχνει διάθεση να συνεργαστεί στον τομέα αυτών. Και γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ζητήσω να πω το εξή ότι η νομιμοποίηση τέτοιων μέτρων για την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών αρχών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αμφισβητείται διαρκώ από του πολίτε. Ε, ε, πρέπει λοιπόν να βρούμε κατάλληλα μέσα και πρότυπα και προδιαγραφέ σε αυτή την αστυνομική και δικαστική συνεργασία. Ευχαριστώ και εκ μέρου του των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών παρακαλώ τον κύριο Τίμωθη Κέρκοπ να λάβει τον λόγο. Πρόεδρε, ως εισηγητής για το EUPNR, για τη συμφωνία δηλαδή περί καταχώρησης των ε, στοιχείων των επιβατών, ε, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει σημαντική ανησυχία ως προς την, ε, από τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται η επιβολή του νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο με τις ύψιστες προδιαγραφές προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών μπορούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Γι' αυτό ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε δύο στόχους με, την, ε, με τις προτάσεις αυτές και την προστασία των πολιτικών δικαιωμάτων αλλά και ένα σύστημα ασφαλούς ανταλλαγή δεδομένων και επιβολής του νόμου. Υπάρχει ανάγκη λοιπόν για ένα τέτοιο σύστημα και θεωρώ ότι μια προσέγγιση που θα ακολουθεί του βασικού κανόνε τη απλή λογική, τη κοινή λογική, θα είναι και πιο ορθή. Και θα ήθελα να καλέσω και του συναδέλφου του Κοινοβουλίου να αναγνωρίσουν ότι δεν μπορεί η οδηγία αυτή να είναι πανάκια και να αντικαταστήσει οτιδήποτε άλλο μέτρο επιβολή του νόμου, είτε υφιστάμενο είτε μελλοντικό. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά μα, πρέπει να συνεχίσουμε τι προσπαθίε μα. Είναι καθήκον μα να προστατεύουμε του Ευρωπαίου πολίτε. Εκ μέρους της ομάδας της Ενωτικής Αριστεράς. Το λόγο έχει η κυρία Κορνέλια Ένστ για ένα λεπτό. Κυρίες και κύριοι, απουσία του Συμβουλίου. Φαντάζομαι ότι θα παρακολουθεί από το βίντεο streaming ε, το, ε, της συνεδρίας του Κοινοβουλίου, αλλά φαίνεται δεν είναι διατεθειμένο συζητήσει μαζί μας. Ε, και θα ήθελα να πω ότι η απουσία του Συμβουλίου από την σημερινή, από την απόψινή συνεδρίαση αποτελεί μεγάλη προσβολή ως προς το κύριο και τη θέση του Κοινοβουλίου. Ε, στο θέμα λοιπόν της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της χρήσης τους ε, στην ε, αστυνομική και δικαστική συνεργασία εμείς απορρίπτουμε τις προτάσεις γιατί έχει καταστεί αυτή η ανταλλαγή των δεδομένων ένα ελντοράντο όχι μόνο με το SWIFT αλλά ένα ελντοράντο ανταλλαγής πληροφοριών στην καθημερινή ζωή και στην παρέμβαση το, στην ζωή των πολιτών. που αξιοποιούνται κατά βούληση, όπως παραδείγματι όταν, ε, όταν ε, διαδηλώνουν οι, οι Ναζί. Έτσι λοιπόν αποθηκεύονται στοιχεία για τους πολίτες και νομίζω ότι είτε πρόκειται για το PNR, είτε πρόκειται για την ε, Europol, είτε πρόκειται για άλλα μέσα θα πρέπει να ισχύουν τα ίδια δεδομένα και οι ίδιες αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το λόγο έχει εξ ονόματος της Επιτροπής η Επίτροπος κυρία Μαρία Δαμανάκη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, I Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για την στήριξη προς τις προτάσεις της Κομισιόν και θα ήθελα να αναφερθώ για ακόμη μια φορά σε δύο κυρία σημεία. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι για την Κομισιόν η πρόοδος σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα σημαίνει ότι θα διαπραγματευτούμε και για, και για τον κανονισμό και για την οδηγία ως πακέτο. Και το, το εννοούμε. Έχουμε ε, δύο νομοθετήματα παρά τη, τα αιτήματα του Κοινοβουλίου. Πρέπει να εστιάσουμε τώρα στην διαδικασία και θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι θα επιμείνουμε σε αυτό. Θα διαπραγματευτούμε και τα δύο νομοθετήματα ως πακέτο. Ένα δεύτερο σημείο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι η νέα νομοθεσία μετά την Λισαβόνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων θα ληφθεί υπόψη. Με αναφορά σε όλες, όλες τις ε, συμφωνίες και τις προτάσεις που είναι συναφείς προς αυτό το θέμα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Πιστεύω, Πρόεδρε, ότι όλοι κατανοείτε ότι πρόκειται περί ενός μείζων σημασίας θέματος. Αναφέρεται σε ανθρωπινά δικαιώματα. Αναφέρεται στις θεμελιώδεις αρχές που βρίσκονται στις συνθήκες και με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα πρέπει να καθοδηγούν τις αποφάσεις μας. Γνωρίζω ότι υπάρχει κάποιο εμπόδιο, θα θέλαμε να το ε, ξεπεράσουμε. Η Κομισιόν βρίσκεται εδώ και είναι τεθειμένη να συνεργαστεί για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες τόσο με το Συμβούλιο όσο και με το Κοινοβούλιο. Και φυσικά καλωσορίζουμε οποιαδήποτε πρωτοβουλία από πλευρά Ιρλανδική Προεδρία, εάν η Ιρλανδική ε, Προεδρία εκ μέρου του Συμβουλίου θα ήθελε να ξεπλοκάρει την κατάσταση. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Επίτροπε. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση κηρύσσεται περιομένη. Το επόμενο συζή... ε, σημείο τη σημερινή διάταξη είναι κοινή συζήτηση σχετικά με την αλληλευτική πολιτική. Εκφωνώ τα νόματα των ε, εισηγητών, έκθεση του κυρίου Κρομπάρτσικ, έκθεση του κυρίου Γκάλαχερ, έκθεση της κυρίας Πατράο Νέβες, έκθεση του κυρίου Φερέιρα και έκθεση της κυρίας Λόβιν. Το λόγο έχει οι πρώτα εισηγητές, ε, καλώ βήμα, τον κύριο Μάρικ Γιώζεφ ε, Κρομπάρσικ για τέσσερα λεπτά.